η ανασυγκρότηση τη οικονομία Υπάρχει ένα πρόγραμμα χρηματοδότηση, το οποίο διαμορφώθηκε και το οποίο έχει συνέπειε επί του προπολογισμού. Όχι όσον αφορά τις ε, πιστώσεις υποχρεώσεων, αλλά έχει υποχρεώσει όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα των εκταμιεύσεων. Δηλαδή, θα πρέπει να υπάρξει επιτάχυνση ε, της ε, εκταμείευσης πόρων υπέρ της Ελλάδος, δηλαδή το 5% όσον αφορά τις διαρροτικές πιστώσεις, αυτά θα πρέπει να εκταμιευθούν ε, αμεληθεί και από την άλλη μεριά όσον αφορά την συγχρηματοδότηση θα έχουμε εντυπωσιακή τέτοια χρηματοδότηση γιατί η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι 100% από πλέον δεν πρόκειται για συγχρηματοδότηση αλλά πρόκειται για χρηματοδότηση αποκλειστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, όσον αφορά τα προγράμματα και τις αναλυθήσει δεσμεύσεις, πρόκειται να γίνουν εκταμιεύσεις ταχύτερα όσον αφορά τις προκαταβολές σχετικές με την προχρηματοδότηση. Η Επιτροπή Ρέτζι είναι η επί σε αρμοδία και σήμερα το πρωί αποφάσισε δυνάμει του άρθρου 50 να ε, υποβάλει έκθεση απλουστευμένη και αυτό για να μην υπάρξει καμία καθυστέρηση για την λήψη των αποφάσεων. Και θα ακολουθήσει ψήφιση από το Κοινοβούλιο κατόπιν. Έχουμε την σημερινή συνεδρίαση των συντονιστών. Το πρωί έγινε για αυτό το θέμα και συμφωνήθηκε να μην γίνει έκθεση γνωμότηση, αλλά μια απλή επιστολή να συνταχθεί αυτή και να την υπογράψει ο πρόεδρος τη επιτροπή σα Και στην Επιτροπή αυτή θα ζητήσουμε από την ε, Επιτροπή κάποιες ε, ε, διευκρινήσεις για τις πληρωμές αυτές. Πρόκειται να γίνει ένας τριμερής διάλογος το φθινόπωρο όσον αφορά τις σχετικές προθεσμίες και είπαμε ότι θα πρέπει να δούμε έγινε, έγινε το φθινόπωρο αυτός ο τριμερής διάλογος και πότε θα πρέπει να δούμε το πώς θα έχουμε την διάρθρωση αυτών των δράσεων. Είναι εδώ ο κύριος Φέζα, μήπως θα μπορούσατε να μας πείτε με λίγα λόγια, να μας πείτε ποιες είναι οι συντρέχουσες βασικές διατάξεις που προβλέπονται από πλευρά ε, κομισιών και ακριβώς ποιες θα είναι οι μέλουσες επιπτώσεις. Κύριε Διευθυντά, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θυμίζω ότι στις 17 εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε μια τροποποιητική πρόταση. Αν δεν έχετε αντίληψη να σα τα πω στα αγγλικά για το κείμενο μου, έτσι θα Άρα μιλάμε για τι 17 Ιουλίου, οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέβασε μια πρόταση σε σχέση με κάποια στροπλήσεις των κοινών διατάξεων για αυτά τα διαφορετικά ταμεία, τόσο ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα σοβαρά προβλήματα χρηματοοικονομικών ροών της ε, Ελλάδας, γιατί μια κατάσταση ήταν τόσο δραματική. Οπότε, ε, με λίγα λόγια, ποιες είναι οι προτινόμενες από εμά ε, αλλαγές. Πρώτα-πρώτα, όσον αφορά το πρόγραμμα του 2014-2020 και σε σχέση με την προηγουμένη προγραμματική περίοδο, περίοδο προγραμματισμού τέλο πάντων, από το 7 μέχρι το 14. Για τα νέα προγράμματα η πρότασή μας αφορά την αύξηση του βαθμού συγχρηματοδότησης ή προχρηματοδότησης όσον αφορά την συνολική διάθεση πόρων για την Ελλάδα. Αυτή την 7 αιτία μιλούμε για ποσό 14,6 δις για την περίοδο αυτή. Οπότε θα γίνει η αύξηση της προχρηματοδότησης κατά 7% και το αποτέλεσμα θα γίνει front-loading αυτών των πληρωμών, γιατί εάν δεν γινόταν αυτή η αλλαγή, θα υπήρχε κατανομή των πόρων στην προγραμματική περίοδο. Όμως ε, ε, αυτού του είδους η μέθοδος θα μας οδηγήσει σε ένα δις και έχουμε 500 εκατομμύρια το 15 και το άλλο μισό, τα άλλα 500 το 16. Επίσης υπάρχει άλλη μια διάταξη στις προκεινόμενες διατάξεις ότι για να έχουμε κάπως μια ταχύ εφαρμογή γιατί είπαμε ότι υπάρχει κίνητρο σοβαρό να έχουμε επενδύσεις να υπάρχουν συνθήκες ώστε η ελληνική οικονομία να μπορέσει να ξαναμπεί στο δρόμο της απασχόλησης και της ανάπτυξης οπότε η σχετική τασόμενη προϋπόθεση είναι ότι για να γίνει η προχρηματοδότηση θα πρέπει να έχουμε για κάποιο είδου αξιώσει πληρωμών και επιστροφών, ούτω ώστε θα πρέπει αυτέ οι αξιώσει να έχουν ληφθεί από την Επιτροπή μέχρι τέλο του 2016. Άλλο, το κομμάτι τη προχρηματοδότηση που δεν θα καλυφθεί από αυτέ τι αξιώσει θα πρέπει να επιστραφεί. Επομένω, ή να ανακτηθεί τέλο πάντων. Αυτό δεν είναι κύρωση, αλλά είναι για να δώσουμε όσο γίνεται πιο ισχυρά κίνητρα, ούτω ώστε να ε, έχουμε κάποιες επενδύσεις στην ελληνική οικονομία. Αυτά όσον αφορά την τρέξω περίοδο προγραμματισμού. Επίσης έχουμε κατεβάσει και άλλες δύο τροποποιητικέ προτάσεις για την προηγουμένη περίοδο προγραμματισμού. Πρώτα-πρώτα έχουμε την αποδέσμευση την προηγουμένη για το 15 σύμφωνα με την προτινόμενη τροποποίηση της νομοθεσίας που αφορά το τελικό 5% το οποίο πρέπει να εκταμιευθεί για κάποιες αξιώσεις του, της περίοδου 7 έως 13, τα σχετικά προγράμματα. Και οι ισχύουσε τώρα διατάξεις προβλέπουν ότι αυτό το 5% το οποίο αφορά όλη αυτή την επταετία πρόκειται να εκταμιευθεί μόνο μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων και λόγω των διαφορετικών κινήσεων που θα πρέπει να γίνουν για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων αυτό το 5% δεν θα εκτομιγόταν πριν το 2017. Αλλά σύμφωνα με την τροποποίηση θέλουμε να κάνουμε κάποια εξαίρεση αυτών των κανόνων των κοινών διατάξεων και θα δοθεί δυνατότητα, θα υπάρχει δυνατότητα αυτό το 5% να εκταμιευθεί από το 2015. Οπότε έτσι θα υπολογιστεί αυτό για την περίοδο 2007 έως 2013. Η δεύτερη τροποποίηση των διατάξεων είναι αυτό που ανέφερε προηγουμένως ο κύριος Πρόεδρος, ότι δηλαδή η χρηματοδότηση αυτού του προγράμματος πρόκειται να ε, καλυφθεί 100% από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, χρηματοδότηση 100% από την Ένωση. Οι δε ε, επιπτώσεις αυτών των δύο τροποποιήσεων επί των προγραμμάτων 2007 2020 είναι ένα ακόμα δις εμπροστοβαρών πληρωμών που θα καταβληθούν 15-16 και όχι αργότερα μέσα στην ίδια περίοδο. Και για αυτό το δις είπαμε ότι το μισό θα αφορά το 15, τον προπολισμό του 2015 και τα άλλα 500 εκατομμύρια θα καλυφθούν από τον προπολογισμό του 2016. Αν τώρα δείτε συνολικά αυτέ τι τροποποιήσει, θα διαπιστώσετε ότι από πλευρά παρόν ρύθμιση έχουμε ένα εκατομμύριο παραπάνω όσον αφορά τις πιστώσει πληρωμών. In 20... Ε, Και επίση το 16. Άρα, το θέμα είναι η κάλυψη πώς θα γίνει όσον αφορά τις εγκριθήσεις ε, πιστώσεις πληρωμών του 2015 και σε σχέση με την πρόταση του Κομισιόν για το 2016. Ένα νέο στοιχείο τώρα το οποίο εμφανίζεται όσον αφορά τον υπολογισμό ε, των αναγκών που θα από τις πληρωμές είναι οι προβλέψεις των κρατών μελών και είπαμε ότι θα πρέπει μέχρι τέλος Ιουλίου να είχαν φτάσει στην Κομισιόν. Η πρόβλεψη ήταν το πόσες αξιώσεις θα υποβληθούν φέτος και του χρόνου. Ακόμα δεν έχουμε λάβει όλες αυτές τις ε, προβολές, τις προβλέψεις. Ακόμα λείπουν πολλές. Πάντως, για το 2015, οπότε παραδοσιακά οι προβλέψεις είναι περισσότερο ακριβείς, τα κρατημέλη δηλαδή ακριβέστερα προβλέπουν το τι αξιώσεις θα υποβάλουν για το τρέχον έτος, δηλαδή το 15 υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις όσον αφορά τα προγράμματα. Και οι αξιώσεις των κρατών μελών είναι λιγότερες από τις προβλέψεις. Οπότε η δική μας εκτίμηση ότι δεν έχουν αυτές είναι ότι έτσι θα μπορέσουμε να καλύψουμε αυτό το έξτρα δισεκατομμύριο για το 2015. Άρα δεν χρειάζεται να αυξηθούν οι πιστώσεις πληρωμών για το 2015. Το 2016. Εδώ δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι 100% γιατί ο βαθμός ακριβίας των προβλέψεων των κρατών μελών για την επομένη χρονιά συνήθως ε, σε σχέση με την πρόβληση ε, του τρέχοντος έτους. Άρα πάμε για ε, αξιολόγηση του 11%. Αυτό είναι σημαντικό και επομένως αυτά που θέλω να σας πω σαν ενδείξεις δεν πρέπει να τα παίρνετε και τη μετρητής. Αλλά αυτό οφείλεται το ότι έχουν μειωθεί οι προβλέψεις κάποιων κρατομέλων για το 2016. Όπως φαίνεται θα μπορέσουμε να καλέψουμε και αυτό το άλλο δισεκατομμύριο όπως προκύπτει από αυτόν τον τροποποιημένο ε, κανονισμό. δεν θα χρειαστεί να αυξήσουμε τις πιστώσεις πληρωμών. Οπότε δεν θα πειράξουμε ότι συμφωνήθηκε ως ε, πρόγραμμα πληρωμών. Επομένως όλα αυτά συνάδουν με το στόχο που είχε ταχθεί, δηλαδή να έχουμε μια, ε, μια, μια, ένα ποσό 20 δις τέλος του έτους που θα ήταν αυτές οι πληρωμές που ακόμα δεν είχαν καταβληθεί. Και επίσης είπαμε ότι έχουμε αυτές τις πληρωμές ε, που δεν έχουν καταβληθεί με τέλος του 2016. Επομένως, αυτές είναι οι προβλέψεις για τα ανεξόφλητα που έχουμε σε αυτή την φάση και αν έχετε συγκεκριμένες ερωτήσεις, πρόθυμα να τις απαντήσω, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Φρέζα για τις διευκρινήσεις αυτές και ένα καλό νέο λοιπόν, μια καλή είδηση δεν θα επηρεάσει τον προγραμματισμό των πληρωμών στο συνολό του, αλλά το κακό νέο είναι ότι ορισμένες αναλήψεις υποχρεώσεων θα αναβληθούν χρονικά οπότε ακριβώς τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να ενθαρρύνει τις επενδύσεις υπάρχει ένας κίνδυνος ε, ε αντίθετης κίνησης ε, ναι, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συναδελφοί, η συμφωνία με την Ελλάδα είναι τόσο σημαντική που μας χαροποίησε και μπορούμε επί της αρχής να συμφωνήσουμε, αλλά θα πρέπει να μας δοθούν κάποιες εξηγήσει. Και έχετε δίκιο στην επιστολή σας που λέτε ότι αυτές οι θέσεις είναι απαραίτητες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι σίγουρα θα υπάρξουν συνέπειες, όπως είπατε, στις πιστώσεις πληρωμών, για τις οποίες υπάρχουν ήδη δυσκολίες. Οπότε αυτό θα πρέπει να παροτρύνει το Συμβούλιο να αφήσει λίγο περισσότερο περιθώριο για το ζήτημα αυτό των πιστώσεων πληρωμών. Αλλά ενδεχομένως, ας το ελπίσουμε, αυτό θα μπορούσε στο μέλλον να βελτιώσει τη διαχείριση των διαρθρωτικών ταμείων για το σύνολο των χωρών, επιταχύνοντα διαδικασίε, γιατί όπω γνωρίζετε σήμερα η μεγάλη δυσκολία στα διαρθρωτικά ταμεία όσον αφορά τι χώρε, είναι οι καθυστερήσει των πληρωμών. Οπότε μπορούμε να φανταστούμε ότι αυτή η εμπειρία θα βοηθήσει τις μεταφορές κονδυλίων στις διαφορές χώρες στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων. Ίσως αυτό λοιπόν είναι κάτι που θα πρέπει να επισημάνετε στην επιστολή σας. Είναι σημαντικό. Σίγουρα θα έχει συνέπειες, αλλά μπορεί να έχει και καλά αποτελέσματα. Ευχαριστούμε. Δεν θα ήταν κακό να είστε σύντομοι συνάδελφοι, γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε στις 6, κύριε Φερνάντες. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος. Ε, φυσικά και ε, Συμφωνώ και χαίρομαι για τη συμφωνία που επιτεύχθη τόσο για τη συγχρηματοδότηση του 100% όσο και για την προχρηματοδότηση από το 2014 μέχρι το 2020. Ε, εδώ μιλάμε για ποσό σχεδόν 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ορισμένα είναι προχρηματοδότηση και σε άλλες περιπτώσεις ε, ε, απαιτούν λιγότερα ε, από την Ελλάδα, οπότε ελπίζω η Ελλάδα να ε, επιτύχει την σταθερότητα αυτή που θα της επιτρέψει να αξιοποιήσει αυτά τα έργα στο μέγιστο. Η αιρεσιμότητα είναι κίνητρο σε τελική ανάλυση. Ενθαρρύνει τη χώρα να χρησιμοποιήσει σωστά τα χρήματα. Αν αυτά τα χρήματα δεν χρησιμοποιηθούν, δεν ε, θα υπάρξουν δεν θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τα χρήματα. Είναι περίεργη η ρεσιμότητα. Αλλά ξέρετε όλοι οι προπολογισμοί είναι μια άσκηση ε, προβλέψεων επίσης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τις συνέπειες όλων αυτών και να μεριμνήσουμε οι διάφορες στρατηγικές να μην ε, επηρεάσουν αρνητικά τα αποτελέσματα των προγραμμάτων. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε γιατί ε, δεν πρέπει να δημιουργούμε προβλήματα ενώ προσπαθούμε να διορθώσουμε ένα και δυστυχώς το Συμβουλίο έχει αυτή τη συνήθεια απλά θέλει περικοπές όλη την ώρα. Τώρα λέει ότι περικόπτει από την μια πλευρά τα κονδύλια και μετά λέει ότι περικόπτει από αλλού και τα βάζει αλλού και έτσι όλα αυτά έχουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Ε, θυμάμαι μια ζήτηση στο ΕΦΣΙ όταν εγώ είχα πει στο Συμβούλιο ότι το να βγάζουμε ένα ευρώ από τη μια τσέπη και να το βάζουμε στην άλλη δεν ε, μετατρέπει το ευρώ σε δύο, εξακολουθεί να είναι ένα. Οπότε να το βγάζουμε από το ένα μέρος και να το βάζουμε αλλού δεν έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Οπότε ε, είναι σημαντικό που το προτείνει αυτό η Επιτροπή. Το να έχουμε ένα buffer φυσικά είναι καλό για τα προγράμματα, διότι ακόμα και αν δεν γνωρίζουμε τι θα ζητήσει το Συμβούλιο από τα κράτη-μέλη όσον αφορά τα εθνικά επιχειρησιακά προγράμματα, τουλάχιστον γνωρίζουμε ότι θα έχουμε ένα πρόβλημα. Έχουμε 20 δισεκατομμύρια ευρώ απλήρωτα το 2015 Έχουμε το στόχο αυτού του 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2017 που μεταφέρεται από το 2007-2013 οπότε έχουμε ένα πρόβλημα για την περίοδο του 2014 μέχρι το 2020 οπότε εδώ είναι σαφές ότι βρισκόμαστε σε μια θέση όπου πρέπει να επιβαρύνουμε όπου επιβαρύνει την κατάσταση οπότε χρειάζεται μια λύση πρέπει να λάβουμε μια πρόταση της Κομισιόν όσον αφορά την στρατηγική που θα υιοθετήσουμε ώστε να μην επιδεινωθεί ε, η καταστάση των προγραμμάτων. Αυτή είναι η αλληλεγγύη που θέλουμε να προσφέρουμε στην Ελλάδα, αλλά δεν πρέπει να βλάψει άλλα επιχειρησιακά προγράμματα σε εθνικό επίπεδο. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ο κύριος Κόλμελ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον εκπρόσωπο για την εκτενή παρουσίαση και για τα τεχνικά διοικητικά που μας εξήγησε. Συμφωνώ με τον προλαλήσατε τον κύριο Φερνάντες. Θέλει προσοχή. Να μην αρχίσουμε να έχουμε ε, μεταφορές κονδυλίων δεξιά και αριστερά. Ε, μία φορά άπαξ καταβάλλονται αυτά. Δεν θα πρέπει να δημιουργούμε αποθεματικά και μετά να πηγαίνω έρχονται τα λεφτά. Όλο και περισσότερο υπάρχει ο πειρασμός ε, να μην λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Γίνεται λόγος για αρνητική ανάπτυξη. Παλαιότερα αυτό το λέγαμε σε ρίκνωση της οικονομίας, ξέρετε. Τώρα μιλάμε για συγχρηματοδότηση, λέει, του 100%. Ωραία ορολογία. Αυτό σημαίνει χρηματοδότηση 100%. Το συν τι το θέλουμε. Άρα να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και όχι τέτοιες ασάφειες γιατί το αξίζουν οι πολίτες ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, για το ίδιο το πρόγραμμα. Και πάλι έχουμε υποκύψει στον πειρασμό. Το λάθος φάρμακο που δώσαμε και δεν επέδρασε, ακριβώς γιατί ήταν λάθος το φάρμακο, τώρα αυξάνουμε τη δόση. Γιατί το λέω αυτό. Διότι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι στην Ελλάδα έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα και σοβαρό ε, με τις διοικητικές δομές και την κρατική μηχανή. Αυτό το πρόβλημα δεν βελτιώνεται εάν λέμε ότι αυξάνουμε τα κονδύλια για την Ελλάδα. Η διοικητική μηχανή και δομή δεν βελτιώνεται έτσι. Και μεταξύ άλλων ευθύνεται και αυτή για το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν ήταν σε θέση μέχρι τώρα να απορροφήσει απολύτως τα κονδύλια. Δηλαδή προσοχή να μην βγούμε και να λέμε ότι δημιουργούμε ένα πρόγραμμα και προβλέπουμε και κονδύλια και όλα θα πάνε καλά. Εμένα μου λείπει ε, η δομή για μια πραγματική βοήθεια για την Ελλάδα και θα ήμουν πάρα πολύ ευγνώμων αν είχατε να μου δώσετε εδώ μια απάντηση σχετικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, να πω μόνο κάτι. Προβλέπετε να δοθούν στο Κοινοβούλιο εξουσίες παρακολούθησης ε, για να εξασφαλίσουμε ε, ότι η δεσμεύση της Ελλάδας για μεταρρυθμίσεις είναι πραγματικότητα και όχι ρητορική, ότι θα υλοποιούνται δηλαδή. Η κυρία Γουαρδία Σάμπαλ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ήταν επιτυχία αυτό που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μια τροποποίηση λοιπόν ε, για τα διαρθωτικά ταμεία για να βοηθηθεί η Ελλάδα και αυξήθηκε η συγχρηματοδότηση και έφτασε στο 100%. Όλο αυτό είναι επιτυχία και το χαιρετίζω. Κατανοώ ότι από πλευρά δημοσιονομικής για τις πληρωμές, αν δούμε την περίοδο 2014-2020, είναι ουδέτερο ως προς τον υπολογισμό. Αλλά υπόθηκε ε, ότι αφορά ιδίω το 2015 και 2016. Αυτό που δεν μπορώ να καταφέρω να καταλάβω είναι πώ υπολογίσατε ότι το ένα δις μπορούν να το απορροφήσουν ε, απολύτως, ενώ έχουμε 20 δισεκατομμύρια ανεξόφλητους λογαριασμούς. Έχουμε μειώσει λίγο την πίεση του Κοινοβουλίου το καλοκαίρι για αυτό το θέμα, γιατί θέλαμε να προχωρήσουμε στις πολιτικές προτεραιότητες. Άρα τι εξαφανίστηκε το πρόβλημα των 20 δις ανεξόφλητων λογαριασμών. Αλλάζουν οι κανόνες και τώρα βάζουμε λίγο ακόμα λάδι στη φωτιά των ανεξόφλητων λογαριασμών. Πού θα το βρείτε. Έχει την ευκαιρία τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη δικαιολογία ή την πρόφαση για να ξαναφέρει το θέμα των ανεξόφλητων λογαριασμών και να ζητήσει και πάλι να αυξηθεί το επίπεδο των πληρωμών. Για να αποσυμφορηθεί λίγο το 2016 και να φτάσουμε στους όχους μας. Να πληρώνουμε τους λογαριασμούς μας και να συζητάμε και για τον προπολογισμό ε, με όρους πολιτικών προτεραιοτήτων. Ευχαριστώ. Η κυρία Βανά. Ευχαριστώ. Και εξ ονόματος των Πρασίνων θέλω να πω ότι θεωρούμε το πακέτο κάτι πάρα πολύ θετικό, το καλωσορίζουμε και την απλουστευμένη διαδικασία. Σήμερα κάναμε εκτενή συζήτηση, όπως είπατε και εσείς Πρόεδρε στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης και κάποιοι συνάδελφοι είναι παρόντες. Το παρουσίασε στο πακέτο η Επίτροπος η κυρία Κρέτσου, αλλά δεν θα πρέπει να λησμονούμε τη σημασία τώρα αυτής της κίνησης και ε, της δυνατότητας προς το παρόν ε, επενδύσεων. Τα διαρθρωτικά ταμεία ε, ευθύνονται τώρα σε μεγάλο βαθμό και για την κατάσταση στην Ελλάδα. Το ανέφερε και ο Προλαλής ακριβώς αυτό το πακέτο Πολλά κονδύλια, εξ όσο γνωρίζω, είναι, προβλέπονται για την τεχνική υποστήριξη, έτσι, για την τεχνική βοήθεια των διαρθρωτικών επενδύσεων και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Άρα λοιπόν έχουμε και εμείς την ευθύνη μας ως ε, βουλευτές ε, ε, να δράσουμε γρήγορα και να μπούμε στην απλουστευμένη διαδικασία. Χαίρομαι πάρα πολύ και για την επιστολή με τις διευκρινήσεις για τη διαδικασία και για τις ανησυχίες μας ως προς το θέμα της ανάληψης υποχρεώσεων. Χαίρομαι για αυτή τη διαδικασία, την ε, ταχεία και την αποφασιστική για να στείλουμε και ένα μήνυμα στις επικείμενες συζητήσεις στο Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μάνκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είπαμε σε σχέση με την πρόταση της Ευρωπαϊκή Επιτροπής για το 2015 ότι πρόκειται να καλυφθούν όλες οι αναμενόμενες εκταμιεύσεις για την εφαρμογή των νέων προγραμμάτων. Επίσης είπαμε ότι θα κολύψουν επίσης και τα ανεξόφλητα, οπότε τέλος της χρονιάς θα έχουμε 8 ε, δις ανεξόφλητα. Οπότε εγώ θέλω να ρωτήσω το εξή. Με αυτού του είδους την εφαρμογή ε, τα μαντάτα είναι άσχημα για μας. Πρόκειται για ε, η περιμερία στην οποία βρισκόμαστε. Οπότε θα έχουμε κάποιες σπόρους που θα μείνουν να χρησιμοποιείται. Και έτσι θα έχουμε 19 αντί για 20 δισεκατομμύρια ανεξόφλητα. Μαζί. Αυτό, Πρόεδρε, το είπε και η συνάδελφος, σήμερα στην ε, Περιφερειακή Επιτροπή αλλά και στη συνεδρίαση των συντονιστών. Οπότε και σταθήκαμε σε μια σειρά από ζητήματα. Πρώτα-πρώτα θα πρέπει να θεωρήσουμε θετικό το ότι επανενεργοποιήθηκε η Επιτροπή και κατέβασε αυτή την τροποποίηση του κανονισμού. Γιατί τώρα υπάρχει πρόβλημα χρόνου και θεωρώ πολύ θετικό επίσης που η Κοινοβουλική μας Επιτροπή κάλυψε το ζήτημα αυτό και επέλεξε την ε, απλουστευμένη διαδικασία γιατί αυτό το πρόβλημα χρονοδιαγράμματος ε, τι θα σήμαινε ότι αν δεν υπήρχε το συντομότερο έγκληση αυτού του πακέτου με κάποια ε, ασυνέπεια ότι δηλαδή δεν θα είχε τη ρευστότητα που χρειάζεται η Ελλάδα οπότε τελικά διάφορα προγράμματα δεν θα μπορούσαν να τρέξουν προγράμματα τα οποία θα έπρεπε να τρέξουν οπότε να το πρόβλημα όλων αυτών που τώρα τους χρωστάμε λεφτά λόγω των προγραμμάτων. Από την άλλη μεριά θα ήθελα να απαντήσω σε κάποιες παρατηρήσεις που ακούστηκαν. Όντω υπάρχουν κάποια προβλήματα που υπάρχουν όσον αυτά κατά μία. αλλά δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα. Αφορούν το σύνολο των ευρωπαϊκών περιφερειών. Για ρίξτε μια ματιά στο θέμα της ε, απορρόφησης και απορροφητικότητας. Θα δείτε ότι υπάρχουν κάποιες ε, ελληνικές περιφέρειες που δεν είναι σε, στους, στους ουραγούς του πίνακα της απορρόφησης των πιστώσεων. Επομένως, είναι αλήθεια ότι το σύνολο των ευρωπαϊκών περιφερειών χρειάζεται επιγόντως απλούστευση. Χρειάζεται πάρα το να μπορέσουμε να περικόψουμε επιτέλους το χαρτοβασίλειο και την γραφειοκρατία που μπερδεύει τους ε, συναλλασσόμενους και όπως ακούστηκε είναι σωστό επίσης το τελευταίο που θα αναφέρω το σχέδιο του οργανισμού είναι από πλάση προπολογισμού τελείως ουδέτερο. Δεν δημιουργεί δηλαδή επιπλέον δαπάνη που επιβαρύνει τον Και ευχαριστώ. γύρω Τζάνι θα είναι το τελευταίο σου, το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ πιστεύω, αντίθετα από ό,τι λένε οι συναδελφοί μου, ότι δεν είναι καλή ιδέα για δύο λόγους κυρίως. Ο πρώτος λόγος είναι πολιτικός. Μετά από την καταστροφή που έκαναν τα θεσμικά όργανα στην Ελλάδα με το τρίτο σχέδιο διάσωσης, δηλαδή τρία σχέδια διάσωσης, δύο αποτυχημένα μπροστά στα μάτια όλων και το τρίτο το οποίο πιθανότητα θα αποτύχει ξανά διότι κατά την μου δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει τα πραγματικά προβλήματα της Ελλάδας μου φαίνεται ότι εδώ είναι σαν να λέμε ναι εμείς προτείναμε να προτείναμε ένα σχέδιο δακρύζοντας ε, για να δώσουμε κάποια περισσότερα χρήματα. Το δεύτερο είναι ότι πιστεύω δεν θα είναι αποτελεσματικό γιατί, γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ελλάδας, κατά την άποψή μου, έχει ένα όνομα και ονομάζεται ευρώ. Εμείς, αν σήμερα είναι να προβλέπουμε χρήματα για την Ελλάδα, μικρά πλεονεκτήματα μπορούμε να προσφέρουμε σε αυτή τη χώρα ως προκαταβόλες ε, τέτοιων κονδυλίων, όλα αυτά θα χαθούν βία διότι η χώρα αυτή έχει ένα νόμισμα υπερβολικά ισχυρό σε σχέση με την οικονομία της. Μια, ένα νόμισμα το οποίο δεν μπορεί να υποστηρίξει, οπότε εντό εισαγωγικών τα χρήματα αυτά θα πεταχθούν στα σκουπίδια. Οπότε εδώ μιλάμε για προκαταβολές μελλοντικών πληρωμών, αλλά όπως είπαν πολύ σωστά ορισμένοι συνάδελφοι, Σήμερα έχουμε σημαντικά προβλήματα πληρωμών. Τι κάνουμε, παίρνουμε τα χρήματα αυτά, τα δίνουμε ως προκαταβολές και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να καθυστερήσουμε άλλες πληρωμές των διαρθρωτικών ταμείων ή άλλων πραγμάτων που αναμένονται εδώ και καιρό. Στο τέλος του 2015 έχουμε ε, ε, πληρωτή ετοιμολόγια 20 δισεκατομμυρίων ευρώ. Δεν νομίζω λοιπόν ότι σε αυτή την περίπτωση η πρόταση της Κομισιόν είναι καλή. Πάμε να, πάμε να, λύσουμε, το πάμε να λύσουμε το πρόβλημα της Ελλάδας δημιουργώντας ένα άλλο στις πληρωμές ε, του προϋπολογισμού. Και έτσι οι προσπάθειες της Κομισιόν ε, και του Κοινοβουλίου αυτού ε, για τα τιμολόγια θα είναι άκαρπες. Ε, πολλές χώρες, όχι μόνο η Ελλάδα, αναμένουν την πληρωμή αυτών των τιμολογίων και αυτό θα επηρεάσει και τις οικονομίες άλλων κρατών μελών. Αυτή είναι η λογική βάσει της οποίας πιστεύω ότι αυτή η λύση δεν είναι η σωστή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κύριε Φρέζα, πολύ σύντομα παρακαλώ, δεδομένη της γιατί ούτως ή άλλως έχω προβλέψει να συντάξω μια επιστολή βάσει των σχολείων που είπατε, έτσι ώστε η Κομισιόν να μας δώσει διευκρινήσεις. Ε, επιθυμούμε μια επιταχυμένη διαδικασία, επιτυχία αυτού του σχεδίου, ε, επανόρθωση της Ελλάδας, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε σαφώς τι συνέπειες που θα έχουν όλα αυτά όσον αφορά τον προγραμματισμό των πληρωμών και να βεβαιωθούμε ότι δεν θα υπάρξει υπερβολική ζημία προς άλλους πιστωτές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα είμαι σύντομος. Πρώτα απ' όλα μιλάμε για μια προκαταβολή ορισμένων, ε, για μια ε, νωρίτερη πληρωμή ορισμένων, ε, καταβολή ορισμένων πληρωμών για ένα διάστημα, όπως είπαμε. Στην περίπτωση της Ελλάδας, το πρόβλημα που προσπαθούμε να επιλύσουμε είναι ένα πρόβλημα ρευστότητας, όπως υπόθηκε η Ελλάδα δεν είχε ούτε έχει πρόβλημα απορρόφησης ε, για, στα προγράμματα από 2007-2014. Μάλλον η απορρόφηση ήταν γρήγορη διότι προσχέθηκε μεγάλη βοήθεια για να επιταχυνθεί και να βελτιωθεί η διοικητική δομή. Οπότε τα τελευταία χρόνια το πρόβλημα ήταν η ρευστότητα όσον αφορά τη δημοσία χρηματοδότηση. Υπήρχαν προθεσμίες πληρωμών, όλοι το γνωρίζουν και έτσι συσσωρεύτηκαν όλες οι πληρωμές ε, οι οποίες ε, χαρακτηρίζονταν από προθεσμίες και εκεί προστίθεται άλλο ένα στοιχείο το οποίο θα έπρεπε να είχα αναφέρει νωρίτερα ένα νέο στοιχείο ρεσιμότητας ε, όσον αφορά τη ρευστότητα το οποίο εισηχθεί και αφορά τα χρήματα που είναι διαθέσιμα για την προχρηματοδότηση. Στα αγγλικά το ονομάζουμε ring fencing. Χρήματα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τους δικαιοχούς των ταμείων, πουθενά αλλού. Και εκεί το Κοινοβούλιο απέδειξε ήδη, ενέκρινε ένα διατάγμα για να το διασφαλίσουμε αυτό, γιατί δεν συνέβαινε πάντα στο παρελθόν. Όσον αφορά το πώς ε, είναι δυνατόν ε, να, να προσθέτεται 2 δισεκατομμύρια μεταξύ του 2015-2016. Γιατί δεν έχουμε περισσότερα πλήρωτα από αυτό που είχαμε εκτιμήσει. Ο λόγος είναι ότι ουσιαστικά βάσει των προβλέψεων των κρατών μελών διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν καθυστερήσεις σε επίπεδο προγραμματικό ε, καθυστερήσει κάποιων πληρωμών που μεταδίδεται για το 2016 και τα επόμενα έτη αλλά και για τα παλιότερα προγράμματα για ορισμένες χώρες υπάρχει μετάθεση από το 2016 προς το 2017. Όλα αυτά ε, εφόσον αποδεχτούμε τους στόχους που έχουμε, δεχθεί, που έχουμε ορίσει για το σχέδιο πληρωμών. Εμείς εκτιμάμε λοιπόν είναι ότι θα τηρήσουμε τους στόχους του προγράμματος πληρωμών και δεν αποκλείεται το 2015 λόγω των προθεσμιών θα το δούμε όμως αυτό το backlog που έχουμε υπολογίσει των 20 δις να είναι μικρότερο. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι υψηλότερο, αλλά δεν αποκλείται να είναι χαμηλότερο, διότι απλά ένα κομμάτι των ε, αιτήσεων αποζημίωσης θα ε, φτάσουν αργότερα από ό,τι είχε εκτιμηθεί μέχρι στιγμής. Ευχαριστούμε κύριε Φρέζα. Λοιπόν, θα ξαναναφερθούμε σε αυτούς 14 Σεπτεμβρίου. Εκείνη τη στιγμή θα υπογράψω εγώ την επιστολή, οπότε Εκεί θα συζητήσουμε το περιεχόμενο. Περνάω στο επόμενο σημείο. Ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστούμε κύριε Φρέζα. Εγώ ως εισηγητής ε, της γνωμοδότησης ε, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμενο θα ήθελα να σχολιάσω την έκθεση αυτή που παρουσιάζω σε εσάς ε, εδώ υπογραμμίζονται οι γενικές, τα γενικά χαρακτηριστικά του εξαμήνου, οι γενικές κατευθύνσεις, ε, το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τις Στρατηγικές Επενδύσεις που θα αποτελέσει μοχλό για τις ιδιωτικές επενδύσεις, ανταποκρινόμενο απευθείας στις επιθυμίες της Κομισιόν στις 28 Νοεμβρίου του 2014, όπου είχαν οριστεί οι βασικοί μοχλοί για το 2015. Υπογραμμίζω επίσης τις αποφάσεις που ελήφθησαν για τη μεταφορά των ιστοσεων ανάληψη υποχρεώσεων ε, που απέμενα από την περίοδο 2017-2013 και μετά την προχρηματοδότηση για την τόνωση της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για τους νέους. Και όλοι γνωρίζουμε σε ποιο βαθμό είναι επίγον το ζήτημα αυτό, το να προσφέρουμε κάποιες προοπτικές στη νεολαία, λαμβάνοντας υπόψη την έκταση της ανεργίας μεταξύ των νέων. Έτσι λοιπόν ε, ε, με ε, την ευκαιρία αυτής της έκθεσης θα προσπαθήσω να υπογραμμίσω σε ποιο βαθμό η έκθεση των πέντε προέδρων όσον αφορά την, οικονομική, Ευρωπαϊκή Οικονομική και Νομισματική Ένωση χρειάζεται έχει μεν καλές προτάσεις αλλά χρειάζεται επιγόντως ε, να επιταχύνει τις προθεσμίες. Πέραν λοιπόν αυτή τη εκθέση, αυτό ε, είναι ένα τρόπο για να επιμείνουμε στα όσα συζητήσαμε σήμερα το πρωί μεταξύ συντονιστών. Ε, μια, έναν προβληματισμό, μια συζήτηση για το ποιο θα μπορούσε να είναι το δημοσιονομικό και φορολογικό πλαίσιο της ε, Ευρωζώνης. Να υπενθυμίσω ότι οι συντακτέ αυτή τη έκθεσης αναφέρθηκαν σε ένα μηχανισμό δημοσιονομική σταθερότητα για την Ευρωζώνη. Τι σημαίνει αυτό. πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό το ζήτημα και να ξεκινήσουμε τη συζήτηση αυτή στο Κοινοβούλιο ώστε να μην αναλάβει την πρωτοβουλία μόνο το Συμβούλιο. Χαιρετίζω την εθέτηση του κανονισμού που εγκαθιδρύει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, υπογραμμίζοντας το ρόλο που διαδραμάτισε το Κοινοβούλιο, ώστε να ελαχιστοποιηθεί και ήταν οξύμορο αυτό, όπως το ανέφερε ο Χωσέ Μανώνε Φερνάντες, να ελαχιστοποιηθεί η μέγιστη επιρροή της χρηματοδότησης του ΕΦΣΥ. Προσπάθησα σε αυτή την έκθεση να είμαι όσο το δυνατόν πιο σύντομος, όπου, τόσο γραπτά όσο και προφορικά. Όποιος επιθυμεί να λάβει το λόγο, να υπενθυμίσω ότι έχουμε στο χρονοδιαγραμμά μας 10 ε, Σεπτεμβρίου για υποβολή τροπολογιών και ότι θα εξετάσουμε τις τροπολογίες ε, και θα ψηφίσουμε στις 30 Σεπτεμβρίου. Η αρμόδια της ουσίας Επιτροπή ΕΚΟΝ θα αποφασίσει 13 Οκτωβρίου και κατά την τρίτη ε, μετρώντας από τώρα ολομέλεια, την δεύτερη ολομέλεια του Οκτωβρίου θα την τρίτη ολομέλεια του Οκτωβρίου θα ε, αποφασίσει για το Ευρωπαϊκό Εξάμενο. Δεν βλέπω να υπάρχουν σχόλια. Περνάω στο επόμενο σημείο και δίνω το λόγο στον Hans για το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση ε, για την υπόθεση Opel από ό,τι βλέπω λιγοστεύουμε συνέχεια και σε κάθε σημείο το συζητάμε ακόμα λιγότερο. Και αυτό και εγώ θα είμαι να σα εξηγήσω αυτή την καινούργια υπόθεση όσον αφορά το Ταμείο με την Παγκοσμιοποίηση. Είναι και εδώ ένα καινούργιο θέμα που επίση έχει να κάνει με την αυτοκινητοβιομηχανία και σα πενθυμίζω ότι πριν από λίγο καιρό είδαμε συγκεκριμένα πάλι το τι γίνεται με την ε, εταιρεία Opel εδώ, στο Βέλγιο, στην Αμβέρσα. Και όλοι ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι οι το και στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω τη ε, κρίση έχουν συρρυκνωθεί και όσον αφορά την περίπτωση τη Opel έχουμε 39% μείωση. Και όταν ε, μιλούμε για το μπόχον που είναι η έδρα της εταιρείας εκεί έχουμε 55% μείωση. Οπότε βλέπουμε ότι αυτό οδήγησε σε απασχόληση 2.800, μείωση απολύσεις των περίπου τα 2.881 άτομα και έτσι γι' αυτό και απευθύνθηκαν οι γερμανικές αρχές του Ταμείου Προσαρμογής και ζήτησαν, αν θυμάμαι καλά, κάτι παραπάνω από 11 εκατομμύρια ευρώ. Με αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα χρηματοδοτήσει κατά ένα 60% δηλαδή 6,9% οπότε έτσι καλύπτονται όλα τα δέοντα και οπότε γι' αυτό ο κύριος Γκάιερ έφτιαξε ε, τη σχετική έκθεση και θα την παρουσιάσει για την ε, στην Επιτροπή των για συζήτηση κλπ. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Η ε, κυρία Βάνα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα λίγο να συμπληρώσω γιατί είμαι μέλος της ομάδας εργασίας στην Επιτροπή Απασχόλησης για το Ταμείο παγκοσμιοποίηση. Είναι και αυτή μια περίπτωση που μας απασχόλησε όπως και στο ε, παρελθόν το Άλιο Σολάρ για να δούμε αν τα κονδύλια που μπορούν να απελευθερωθούν από εκεί ε, να μην αντικαθιστούν κάποιες υποχρεώσεις και κάποια μέτρα των κρατών μελών. Γιατί αυτό δεν γίνεται με βάση ε, την κοινοτική νομοθεσία. Και στην προηγούμενη υπόθεση ε, δεν μπορεί αυτό να χρησιμοποιηθεί για να ξεπλύνει από τις ευθύνες του τα κράτη-μέλη ε, για τις υποχρεώσεις του απέναντι στους ανέργους κτλ. Ε, και εμείς οι πράσινοι έχουμε τις επιφυλάξεις μας ε, ως προς την νόμιμη ε, χρήση αυτών των πόρων. Ευχαριστώ. Δεν θέλει κανείς άλλο το λόγο. Οι τροπολογίες θα πρέπει να κατατεθούν το αργότερο στις 15 Σεπτεμβρίου. Η Επιτροπή θα το συζητήσει, θα το εξτάσει και θα το ψηφίσει στις 30 Σεπτεμβρίου. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Φερνάντες ο οποίο αντικαθιστά τον κύριο Ρούμπιχ για μια δεύτερη έκθεση για το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση με θέμα τη Ford αυτή τη φορά. Στην Γκένκ εδώ στο Βέλγιο. Ford Γκένκ. Όχι Τζένκ, Γκένκ λέει ο κύριο ε, Ντεπρέ. Ε, καλά, <laughs> εντάξει. Γκένκ, ε, Χένκ κανονικά είναι. Je vou apresentar o relatório em nome do meu Rubik. Λοιπόν, εξ ονόματος του συναδέλφου μου του Πολουρούμπικ θα παρουσιάσω αυτήν την ε, έκθεση. Πρόκειται για μια ερώτηση που αφορά το θέμα των ανέργων που εργάζονταν σε 12 εγκαταστάσεις που επλέξαν από αυτό το μέτρο των ε, 4.881 απολύσεων. Ο συνολικός απολογισμός είναι 10 εκατομμύρια ευρώ. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι, η συμβολή του EGF είναι 6.268.564 ευρώ. Εφόσον δεν υπάρχουν λοιπόν προβλήματα, εμείς είμαστε υπέρ αυτής της κινητοποίησης του Ευρωπαϊκού ε, Ταμείου Προσαρμογής την παγκοσμιοποίηση ώστε να βοηθήσουμε τον καθένα από αυτούς τους ανθρώπους που βρέθηκαν άνεργοι ε, λόγω της παγκοσμιοποίησης για, τη, για αυτό το σκοπό έχει δημιουργηθεί αυτό το ταμείο. Ευχαριστούμε κύριε Ισηγητά. Εδώ υπάρχουν παρατηρήσεις. Κύριε Ντεπρέ. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι σκιώδης συζητητής ε, της Άλντε για αυτό το φάκελο. Μια διευκρίνηση πρώτα απ' όλα. Αναφερθήκατε στην Γκένκ ε, και εγώ σας έκανα παρατήρηση γιατί η Χένκ είναι μια φλαμαδική πώληση, ε, πόλη, συγγνώμη, και στα φλαμαδικά το G προφέρεται Χ, Χένκα. Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Φερνάνδης μου παρουσίασε το... Κύριε Φερνάνδης, είναι πρωτεύουσα σημασίας. Ε, έκανε, είχε μεγάλη, επί, ε, μεγάλη επίδραση στην περιοχή αυτή του Βελγίου όπου υπάρχει ισχυρή αυτοκινητοβιομηχανία και όπου με τη σημερινή ε, μεγάλη παραγωγή που έχουμε στην Ευρώπη Τότε με τη διεύθυνση της ΦΟΡΤ και το προσωπικό είχε καταλήξει σε μια επίσημη συμφωνία υπογεγραμμένη και από τα δύο μέρη που διασφάλιζε την απασχόληση μέχρι το 2020 και τον Αύγουστο του 2012 η διεύθυνση βεβαιώνει ότι θα διατηρήσει τις θέσεις μέχρι το 2020 και τον Οκτώβριο ανακοινώνει το κλείσιμο της επιχείρησης. Με μια σκληρότητα εντυπωσιακή σε μια περιοχή που δεν είναι και η πιο βιομηχανοποιημένη του Βελγίου, οδήγησε 4.000 άτομα στην ανεργία και όλους τους υπεργολάβους που, ε, τους οποίους, οι οποίοι συνεργάζονταν, τεράστια αύξηση της ανεργίας στην περιοχή, σημαντική απώλεια της οικονομικής δραστηριότητας η οποία έπεσε κατά περισσότερα από δύο σημεία το για το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της περιοχής ε, και ε, ανεργία σε μια περιοχή που δεν είναι, όπως είπε και η πιο εκβιομηχανισμένη του Βελγίου. Δεδομένου του αριθμού των ατόμων και των συνθήκων υπό τον οποίο ε, παρουσιάστηκε αυτό το πρόβλημα και χαιρετίζω μάλιστα τον συναδελφό μου τον Κατία Σαμπάλ, διότι η παραγωγή της ΧΕΝΚ ε, μεταφέρθηκε στην Βαλένθια. Οπότε ήδη βίωσα μια αλληλεγγύη από όλες τις χώρες της Μεσογείου και τον Χωσέ Φερνάντες ναι, ε, ε, το νιώσαμε ότι ήταν ε, πολύ αποφασισμένος ο εισηγητής. Ωραία, λοιπόν, ευχαριστούμε για αυτή την έκκληση. Είχαμε πιστεί ήδη, αλλά τώρα ανυπομονούμε να ψηφίσουμε. Τελευταίος ομιλητής, Αντρέι Νοβάκοφ, για την έκθεση του Ταμείου Αλληλεγγύης ε, για τις καταστροφές στη Βουλγαρία και στην Ελλάδα το 2015. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Συνήθως ε, λένε Vox Populi, Vox Dei. Φωνή λαού, φωνή Θεού λέγανε παλιά, ή και οργή Θεού. Σήμερα φαίνεται δεν ακούμε πάρα πολύ τη φωνή του λαού, αλλά του Θεού. Και τελικά, Ευρώπη δεν είναι μόνο ύμνος στη χαρά ή η σημαία ή ξέρω κάποια κείμενα κανονισμών οδηγιών τελικά η ουσία της Ευρώπης είναι η αλληλεγγύη οπότε η αλληλεγγύη όμως θα πρέπει να αποδειχθεί ότι υπάρχει. Και βοήθεια πάνω να πει έγκαιρη βοήθεια. Μιλάμε για 243 εκατομμύρια ευρώ. Ε, σε αυτό το ύψος έχετε η ζημία. Από αυτές τις καταστροφές, τις ε, πλημμύρες, τις κατολιστήσεις κλπ. Καταστράφηκαν ε, παιδικοί σταθμοί, θέατρα, κοινωτικές ε, δομές. Ε, μιλάμε για καταστροφή ανθρωπίνων ζώων και αυτό συνέβη σε πάρα πολύ μεγάλη κλίμακα για κάποιο κράτος το οποίο πολεμάει κατά της 400 εκατομμύρια ευρώ και παραπάνω ήταν καταστροφές στην Ελλάδα και στις δύο χώρες πάνω από 10% των ε, προκαταβολών εκταμιεύτηκαν. Και λέμε ότι στην Ευρώπη έχουμε 50, 15 δραστοδομόσφαινα κράτη και μία ομόσπονη περιοχή. Δηλαδή ο, είναι δυνατόν ο κόσμος έτσι να θεωρηθεί ότι είναι Ευρωπαίοι, να αισθανθούν Ευρωπαίοι. Δηλαδή θα πρέπει να φέρουμε την Ευρώπη κοντά στον ε, πολίτη. Αλλά αυτό να γίνεται και στις αναποδίες και στον καλό γέριο. Και μιλάμε τώρα για αυτές τις θεομηνίες σε Ελλάδα και Βουλγαρία. Και το εξής, οποτεδήποτε υπάρχει μια τέτοια περίσταση θα πρέπει πάντοτε να ενεργούμε με την ίδια μέθοδο. Δηλαδή, μέσα σε ένα εξάμεινο να έχουμε καταβάλει τις σχετικές αποζημιώσεις. Και γνωρίζω ότι δεν προβλέπεται εκτακτή βοήθεια, όμως τα κράτη-μέλη θα πρέπει να καταβάλουν αυτά που οφείλουν εγκαίρως και όταν πρέπει να πληρώσει η Ευρώπη είναι περίμερη, καθυστερεί. Δεν το καταλαβαίνω. Επομένω, συνάδελφοι, γι' αυτό σα λέω, εγκρίνεται αυτή την έκθεση, οπότε έτσι θα μπορέσουμε να δώσουμε τη βοήθεια του συντομότερο δυνατόν και στι δύο χώρε. Στι δύο χώρε που χτυπήθηκαν από αυτέ τι ε, θεομηνίε. Και όταν στο μέλλον υπάρχει μια τέτοια περίπτωση, θα πρέπει πάντοτε να καταβάλλονται οι αποζημιώσει το συντομότερο δυνατόν. Ευχαριστώ κύριε Σεγητά για ε, ε, αυτή σας την ε, στεναρή παρουσίαση και κύριε Φρέιζερ το συντομότερο να γίνει η εκταμείευση και αφού συμφωνούμε όλοι ευχαριστώ πολύ τελειώσαμε τη μερίσια διάταξη δεν έχει κανείς τίποτα άλλο να θέσει να σας πω πότε είναι η επόμενη συνεδρίαση 14 και 15 Σεπτεμβρίου εδώ στις Βρυξέλλες λήξη συνεδρίασης